Οπότε εγκρίνεται ο διορισμός του. Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη τώρα. Το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξης που έγινε δεκτό από την διάσκεψη των Προέδρων στις 9 Δεκεμβρίου δυνάμει του άρθρου 137 του εσωτερικού κανονισμού δημοσιεύτηκε. Για τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν υπάρχει καμία αλλαγή, καμία εισήγηση, καμία... οπότε θα περάσω κατευθείαν στην Τετάρτη. Η ομάδα ΕΛΚ ζήτησε την προσθήκη του κυρίου Σάγερ για τον έλεγχο που διεξάγουν τα κράτη-μέλη ως προς την άσκηση κάποιων αρμοδιοτήτων, εφαρμοστικών ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Σάγερ, σας δίνω το λόγο. Πρόεδρε, όπως είπατε σωστά, ζητούμε να μπει στην μερίσια διάταξη ο κανονισμός για την εφαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων της Επιτροπής και είναι κάπως παράξενο αυτό, δεν είναι έτοιμα μόνο τη ομάδα μου και άλλες ομάδες υποστηρίζουν την ιδέα αυτή και στην νομική επιτροπή υποστηρίχθηκε αυτό. Από όσο έχω καταλάβει υπάρχει ομόφωνη άποψη περί αυτού. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχει πέρασει ένας χρόνος από την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα. Ο κανονισμός αυτός για τις εφαρμοστικές πράξεις είναι κάτι που προέκυψε μετά από ένα χρόνο μακρών διαπραγματεύσεων ε, στον τομέα των ε, ε, στον τομέα αυτό των διατάξεων που είναι πολύ σημαντικός για το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να συζητηθεί και να ο νέος αυτός κανονισμός το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα επίσης να σας πω, Πρόεδρε, όπως ξέρουν και οι συνάδελφοι, ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρχαν δύο ε, αναστέλουσες μειοψηφίε και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησε. Πιστεύω ότι είναι το σωστό να προχωρήσουμε για να κλείσει το θέμα το συντομότερο δυνατό. Ε, τηρούνται όλα τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στην έκθεση αυτή και ζητώ την υποστήριξη και των υπόλοιπων ομάδων ε, ε, στο έτοιμά μου αυτό. Ποιοι είναι υπέρ τη υπέρ της αυτός ο κ. Σφόμποντα. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε αντίρρηση να εγγραφεί στην ημερησία διάταξη. Σημειώνω ότι από ορισμένε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ εξεφράστησαν επιφυλάξει ό,τι αφορά τι συγκεκριμένε ρυθμίσει. Πρώτα, χρειαζόμαστε σίγουρα μια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ώστε το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, μάλλον την Πέμπτη θα μπορούμε να ψηφίσουμε. Ήδη δεν μπορώ να πω εάν είναι δεδομένη η σύμφωνη ή μη σύμφωνη γνώμη μας. Πάντως συμφωνούμε να εγγραφεί στην ημερησία διάταξη. Ε, όλα είναι έτοιμα, ε, λέει ο πρόεδρος Μπούσεκ σε ό,τι αφορά δηλαδή τις προθεσμίες, εφόσον βεβαίως αποβεί θετική η ψηφοφορία. Κατά τις προτάσεις, παρακαλώ, κατά τις προτάσεις. Ποιος θέλει να πει λίγα λόγια. Κανείς. Καλά λοιπόν. Ψήφι υπέρ της προτάσεως. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. για να το εκφράσω ακριβέστερα. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί συζήτηση, την Τετάρτη. Και η συνάντησή μας, η συνεδρίασή μας της Τετάρτης, της Ολομέλειας δηλαδή, θα διαρκέσει μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι τροπολογίες μέχρι Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 10 η ώρα, 10 το πρωί. 10 το πρωί λοιπόν Τετάρτη οι τροπολογίες. Ψήφο την Πέμπτη, ψηφοφορία την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ. Άλλη πρόταση από σοσιαλιστές και δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζήτησαν να υπάρξει προσθήκη μιας ε, προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την οικονομική διακυβέρνηση βάσει και το άρθρο, την λειτουργία του άρθρου 9 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ζητείτε να προσθεθεί αυτό στην ημερήσια διάταξη. Η πρόταση θα υποβληθεί από την κυρία Τρότμαν, εξ ονόματο των Σοσιαλιστών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου όντω θα ήθελε να επανατεθεί προσυζήτηση, να επανατεθούν συζήτηση δύο προφορικές ερωτήσεις για την έκθεση της Task Force και το νομοθετικό πακέτο της Επιτροπής για την Οικονομική Διακυβέρνηση για θεσμικούς λόγους καταρχάς. Το έθνο 9 της Συνθήκης της Λισαβόνας ε, μας δίνει τις εξουσίες και την αρμοδιότητα να μπορέσουμε να ζητήσουμε την, την εφαρμογή της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρε, δηλαδή, ιδιαίτερα τη μελέτη κοινωνικού αντικτύπου για τις μεγάλες αποφάσεις, οδηγίες που έχουν συνέπειες ε, στους πολίτες. Ο κ. Μόγκ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας ε, Συνδικάτων, ε, εξέφρασε γραπτό τις ανησυχίες του για το πρόγραμμα λόγω του προγράμματος λιτότητας σε ό,τι αφορά τους μισθούς των και τη συντάξη των μισθωτών. Ο λόγος για τον οποίο θέτουμε το ερώτημα αυτό, Πρόεδρε, είναι ότι τη στιγμή που συζητούμε την ρύθμιση της αγοράς δεν μπορεί να μην λάβουμε θέση υπέρ της αγοράς αλλά υπέρ των πολιτών μας. Θα ζητούσε λοιπόν από το Σώμα να υποστηρίξει το αίτημα επανυποβολής της προφορικής ερώτησης. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να μιλήσει κατά, ε, ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ της πρότασης αυτής. Ποιος θέλει το λόγο για να υποστηρίξει το αίτημα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακριβώς λόγω των σχέσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Συμβούλιο, Επιτροπής και Κοινοβουλίου, θεωρώ σκόπιμο να υποστηρίξουμε την πρόταση της συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να μιλήσει κατά της προτάσεως αυτής. Ποιος είναι κατά της προτάσεως αυτής. Δεν βλέπω κάποιον. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ της προτάσεως. Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση. Οι δύο προφορικές ερωτήσεις θα προσθεθούν το απόγευμα της Τετάρτης. και η συνεδρία θα κρατήσει μέχρι τις 9 το βράδυ. Η μερίσια διάταξη, εγκρίνεται νομίζω η μερίσια διάταξη γιατί δεν έχει προβλεφθεί καμία αλλαγή για την Πέμπτη. Μπορούμε κατά συνέπεια να θεωρήσουμε ότι η μερίσια διάταξη έχει γίνει δεκτή και προχωρούμε στην ε, έναρξη των εργασιών με τις παρεμβάσεις του ενός λεπτού βάσει του άρθρου 150 του κανονισμού. Uh... Συνάδελφοι, όσοι δεν θέλουν να.